Euh, Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Σας καλωσορίζω στη δημόσια ακρόαση για τους στόχους της χιλιετίας ε, ε, και την ανάπτυξη μετά το 2015 θα συμπροεδρεύσουν οι Τέι Τέιλορ, Μάικολ Κάσπαρ και Φίλι Κάσμαρεκ. Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν το 2000 τους 8 στόχους της χιλιετίας για την ανάπτυξη με στόχο να μειώσουν κατά το ίμιση την ένδια στον κόσμο μέχρι το 2015. Παρά τις κάποιες προέδρους, θα πρέπει να πούμε ότι με κάποιες εξαιρέσεις δεν καταφέραμε να σεβαστούμε αυτούς τους στόχους ε, ε, και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους στοχότερους πληθυσμούς. Οι στόχοι αυτοί δεν είναι ε, επιλογή, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν στην απόλυτη ένδια. Θα πρέπει να επενθυμίσουμε κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ γνωστά. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινούν στον κόσμο και αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο πληθυσμό και γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την αποτυχία. Μία αποτυχία η οποία οφείλεται στην έλλειψη χρηματοδότησης και οφείλεται κυρίως ε, στην έλλειψη συνέπειας της εξωτερικής πολιτικής και δε, στην έλλειψη μέτρων ε, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις παράνομες οικονομικές ροές και τα δημοσιονομικά προβλήματα. η καλή θέληση, όσο βαρύτητη και αν είναι, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε και πολιτική βούληση και θα πρέπει να μπορέσουμε να επανεξετάσουμε μοντέλα και μεθόδους ε, τα οποία έχουν αποτύχει στο παρελθόν. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν για την ακρόαση αυτή και ε, για το γεγονός ότι έχουμε γνωσμένου κύρους ομιλητέ για να μπορέσουμε να δούμε συνολικά το θέμα των στόχων της χιλιετίας μετά το 2015 ε, και όσον αφορά την υλοποίησή του, ε, τον επανακαθαρισμό του ή να δούμε κατά πόσον θα πρέπει να του εγκαταλείψουμε για να αναλάβουμε πιο ε, ε σημαντικές δεσμεύσεις. Να δώσω λοιπόν αμέσω το λόγο στον Τέιλορ, ο οποίος θα προεδρεύσει στο πρώτο πάνελ. Κύριε Τέιλορ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζολή, και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά όλους εσάς εδώ σήμερα για αυτή την τόσο σημαντική συνεδρίαση για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας μετά το 2015. Μια ε, πολύ ευρωπαϊκή δέσμευση. Όπως είπε και η κυρία Ζολή, ο, ο συνάδελφος Κάσμαν και εγώ θα προεδρεύσουμε στο πρώτο τμήμα της ακρόασης και ο κύριος Κάσμαρεκ στο δεύτερο τμήμα έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος προκειμένου να επιτευθούν οι στόχοι της χιλιετία, οι οποίοι συμφωνήθηκαν από τους παγκόσμιους ηγέτε πριν από 10 περίπου χρόνια. Οι κυβερνήσει, τα Ηνωμένα Έθνη και οργανώσει τη κοινωνίας των πολιτών κατέφεραν να σώσουν πολλές ζωές και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης ακόμα περισσότερων. Όπως αναφέρεται στην έκθεση προόδου του 2012 των Ηνωμένων Εθνών για τους στόχους της χιλιοτίας, ο στόχος της μείωσης της απόλυτης ένδυας κατά το ίμιση έχει επιτευχθεί. Όπως επίσης επετεύθηκε ο στόχος της μείωσης του ποσοστού των ανθρώπων που δεν έχουν ε, πρόσβαση ε, σε πόσιμο νερό, σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού. Επίσης, οι συνθήκες διαβίωσης 200 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν ε, βελτιώθηκε και ε, το ποσοστό των κοριτσιών έχει εξισωθεί με το ποσοστό των αγοριών. Επίσης, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο για να μειώσουμε την παιδική και βρεφική θνησιμότητα και τη θνησιμότητα των μητέρων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και επίσης προσπαθούμε να μειώσουμε την, ε, τον ανθρώπινο πόνο και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε τις πρακτικές μας. Το 2015 πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίων ε, θα χρησιμοποιούν ακόμα πηγές νερού οι οποίες δεν έχουν βελτιωθεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα πόσιμο. και ένα δισεκατομμύριο περίπου άνθρωποι θα ζουν με ένα εισόδημα λιγότερο του 1,25 δολαρίου καθημερινώς και θα εξακολουθεί να ε, υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό παιδικής θνησιμότητας. Γυναίκες και παιδιά θα πεθαίνουν από ασθένειες οι οποίες μπορούν να προληφθούν. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, η πείνα εξακολουθεί να είναι μια ακόμα παγκόσμια πρόκληση. Επειδή δεν υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες υγιεινής, ε, πρόοδος ε, στην υγεία και στην καλή διατροφή, ε, υπάρχουν απώλειες στην βιοπικιλότητα και η αύξηση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου και αυτό σημαίνει ότι απειλούνται και οι άνθρωποι και τα οικοσυστήματα. Όπως είπε ο κύριος Μπανκιμούν, η επίτευξη των στόχων της χιλιετίας μέχρι το 2015 αποτελεί μεν πρόκληση, αλλά είναι κάτι που είναι εφικτό και πολλά εξαρτώνται από το κατά πόσον θα επιτευχθούν οι στόχοι του MDG 8, που είναι η ε, παγκόσμια εταιρική σχέση για την ανάπτυξη. Εν καιρό οικονομικής και ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, θα μπορέσουμε είτε να επιταχύνουμε ή να αναστρέψουμε την πρόοδο που έχουμε επιτύχει μέχρι τούδε. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυναμική αυτή για να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία του 2015. Ήγηκε λοιπόν η ώρα να δούμε τι πλαίσιο θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε μετά το 2015 και το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι να εξετάσουμε τι διδάγματα έχουμε αντλήσει από το παρελθόν και τι περιορισμούς έχουμε από το ε, συνεχώς εναλλασσόμενο τοπίο. Όπως ξέρετε υπήρξαν αρκετές διαμαρτυρίες για τους παρόντες στόχους της ηλιετίας. Κάποιοι λένε ότι οι στόχοι ήταν ασυνεπείς, κάποιοι λένε ότι η επίτευξη των στόχων ε, υποκρύπτει γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες και κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι αποτελεί καρικατούρα ε, και ότι οι στόχοι της χιλιατίας ε, ήταν κάτι το οποίο επινόησαν οι πλούσιες χώρες σε μια αίθουσα που αποφάσισαν πώς θέλουν να σπαταλήσουν τα αναπτυξιακά κονδύλια αντί να βοηθήσουν φτωχέ χώρες. Πολλοί λοιπόν θεωρούν ότι οι παρόντες στόχοι της χιλιετίας έχουν σημαντικές ελλείψεις ε, και δεν αξιολογείται καταλήλωση πρόοδος. Ε, βέβαια όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Το Σεπτέμβριο φέτος μια ειδική εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών θα δει τι συνέχεια μπορεί να γίνει στις προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξη των στόχων της ηλετίας και κατά πάσα πιθανότητα θα τεθεί και το ζήτημα του τι μέλη γενέστε μετά το 2015. Μπορεί να φαίνεται λίγο πιο δύσκολο να συμφωνήσουμε τώρα σε νέους στόχους ε, ε, σε σχέση με το 2000, λαμβάνοντας υπόψη και τις ουσιαστικές αλλαγές που είχαμε σε παγκόσμιο, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη στις αναδυόμενες οικονομίες ε, αποτελεί το βασικό μοχλό της παγκόσμιας ανάπτυξης και ταυτόχρονα οι ανισότητες ε, μεταξύ και εντό των αναπτυσσόμενων χωρών έχουν αυξηθεί και το ε, κατακεφαλήνα ΕΠ κάποιων ε, χωρών αναδεόμενων μεσαίου εισοδήματος υπερβαίνει το ΑΕΠ κάποιων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η επισητιστική ασφάλεια, η αύξηση του πληθυσμού της γης, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και η ανεργία αφορούν όλους τους ενδιαφερομένους σε θέματα ανάπτυξης, κυβερνήσεις, ιδρύματα, think tanks, ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και όλοι ε, και όλες αυτές είναι ιδιαίτερα απαιτητικέ προκλήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν συμβιβασμοί από όλες τις πλευρές ε, προκειμένου να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα αντικαταστήσει τους στόχους της χιλιετίας ελπίζουμε το τοπίο μετά το 2015 να μας βοηθήσει να υπερβούμε κάποιες από τις ελλείψεις μας και η προφανής έλλειψη είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ε, αναφορά στην ανισότητα. Όπως σας είπα, το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε κάποια από τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να αντιλήσουμε από τους στόχους της χιλιετίας και να εξετάσουμε και τι περιορισμούς είχαν. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν, ας προχωρήσουμε με το πρόγραμμά μας, αν είστε όλοι άνετα, και να δώσω το λόγο στο συνάδελφο Μάικολ Κάσμαν, προκειμένου να παρουσιάσει το επόμενο τμήμα της συνεδρίασης. Παρακαλώ. Yes, you can uh, applaud if you... Μπορείτε και να χειρακροτήσετε αν επιθυμείτε. Δεν είναι το να ακούει κανεί, αλλά το πραγματικά να καταβάλει προσπάθειε. Ευχαριστώ για τι προσπάθειέ σα. Μάικλ Κάσμαν είναι το όνομά μου. Είμαι επικεφαλή ε, για την ε, αναθεώρηση των στόχων ηλιετία. Δυστυχώ ο επίτροπο Πίμπαξ δεν μπορεί να παραστεί σήμερα το πρωί. Για σοβαρό λόγο που συνδέεται με την οικογένειά του. Του στέλνουμε κάθε καλή επιθυμία για ανάρρωση και σε σχέση με το Γενικό Διευθυντή της ε, ε, ΕΝΚΟ θα δώσω τον λόγο στον Κλάους Ρούντισάουζε για 10 15 λεπτά. Έχεις τον λόγο Κλάους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ συμπρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ζητώ συγγνώμη για την απουσία του Επιτρόπου Πίμπαξ που δεν μπορεί να παραστεί δυστυχώ σήμερα το πρωί ανάμεσά σα. Πολύ θα ήθελε να συμμεριστεί τι αρχικέ σκέψει του για το πολύ σημαντικό θέμα τη σημερινή μα ακρόαση μαζί σα. Πρώτα απ' όλα σα αποστέλει όμω τι καλύτερε ευχέ του. Γι' αυτό το πολύ σημαντικό έτος 2014 λέει ο μιλητής που θα είναι σημαντικό έτος για την πολιτική για την ανάπτυξη. Θα είναι το έτος κατά το οποίο θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση της εφαρμογής ε, της ε, ημερήσιας διάταξης με το θεματολόγιο που πέρυσι παρουσίασε ο Επίτροπος Πίμπαλξ. Θα δούμε, ευελπιστούμε, μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό για τα επόμενα 7 έτη, ιδιαίτερα για τον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη. Όλοι γνωρίζετε, πιστεύω ιδιαίτερα, ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης οι προοπτικές για μια πολύ σημαντική από πλευράς κονδυλίων δράση, από πλευράς των εξωτερικών μας δράσεων, δεν έχει ακόμα ε, εξασφαλιστεί ε, η υποδομή. Και θα ξεκινήσει φέτος ε, και το έργο για τους στόχους της χιλιετίας μετά από την έγκρισή τους. Να θυμόμαστε το 2015 είναι δύο χρόνια ακόμα μακριά μας. Η πρώτη προτεραιότητα και σίγουρα η πρώτη προτεραιότητα του Επιτρόπου Πίμπαρξ να κάνουμε ό,τι μπορούμε ακόμα παραπάνω για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους σημερινούς στόχους της χιλιετίας. Η πρόοδος είναι άνηση και εμβαλωματική κιόλας ακόμα. Και όπως ο κύριος Τέιλορ, Τέιλορ μόλις ε, εξέθεσε, πολλά πράγματα απομένουν να γίνουν. Ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς όπου η πρόοδος είναι πολύ βραδία, ιδιαίτερα για κάποιες ευάλωτες χώρες, κάποια ευάλωτα κράτη. Προσπαθήσαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, μεταξύ άλλων με, την, ε, το θεματολόγιο για τις αλλαγές, να χαρτογραφήσουμε πώς θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την επιρροή μας, την επιρροή των κονδυλίων για την ανάπτυξη, ακριβώς για να επιταχυνθεί η διαδικασία προσεγγίζοντας ε, προς την προσπάθεια να προσεγγίσουμε τους στόχους της χιλιετίας και σε σχέση με τα κονδύλια, ένα δι για παράδειγμα για του στόχου τη χιλιετία που ξεκίνησε ως πρωτοβουλία πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Τώρα, τούτων λεχθέντων, οι διάφορες διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους που κάναμε και διεξαγάγαμε με αυτό το, για αυτό το θέμα, για την εργασία μας αποκάλυψαν πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει έντονη υποστήριξη για αυτούς τους στόχους της χιλιετίας ως προσέγγιση θα πρέπει να συναγάγουμε τα συμπεράσματα, να δούμε από τα μαθήματα που μάθαμε τι μπορεί να συναχθεί. Είναι μια πιστική προσέγγιση η στόχη, αναπτυξιακή στόχη της χιλιετίας και μπορούν αυτοί οι αναπτυξιακοί στόχοι χιλιετίας να αποτελούν έμπνευση για τη δραστηριότητα, δραστηριοποίησή μας στον τομέα της ανάπτυξης. Τώρα, αυτό και άλλα συμπεράσματα οδήγησαν τον Επίτροπο Πίμπαρξ να κάνει τι να ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για το πλαίσιο μετά το 2015. Ευχάριστα σημείωσε ότι ζητήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κιμούν ο κύριος Πίμπαλξ να είναι μεταξύ εκείνων των υψηλών αξιωματούχων που θα συνεχίσουν, θα αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία και στη Μονρόβια της Λιβερίας. Ξεκινώντας αυτή τη σκιαγράφηση, τι θα μπορούσε να είναι η διαδικασία για τον ορισμό, προσδιορισμό των αναπτυξιακών στόχων συλλιετίας μετά το 2015 άμεση προτεραιότητα να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το δυνατόν γοργότερα αυτές τις αρχές, αλλά να προβληματιστούμε και να δούμε ποιες θα είναι οι αρχές που θα μας εμπνέουν για την αναπτυξιακή μας πολιτική μετά το 2015. Πιστεύω ότι είναι σαφές για όλους ότι δεν είναι μόνο θέμα κονδυλίων. Η αντιμετώπιση και αναχέτηση καταπολέμηση της φτώχειας δεν είναι μόνο θέμα κονδυλίων. Τα χρήματα διαδραματίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Όμως η απουσία έλλειψη υγείας, ε, κατάρτισης, εκπαίδευσης, οικονομικών ευκαιριών, θέσεων εργασίας, απασχόλησης, δικαιοσύνης, δίκαιου, ε, ισοδίκαιου πεδίου δραστηριοποίησης, ασφάλειας, δικαιοσύνης, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν γίνεται λόγος για αυτό το πλαίσιο μετά το 2015 για την ανάπτυξη. Να ενταχθούν τώρα όλα αυτά υπό μια κοινή στέγη ή με μια πρόταση να καλυφθούν Πώς μπορεί να γίνει. Ο Επίτροπος ε, Πίμπαλξ έχει το στόχο να μπορέσουν όλοι να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση μέχρι το 2030. Εκπαίδευση, παιδεία, οικονομικές ευκαιρίες, ε, δικαιοσύνη, ειρήνη, ασφάλεια, δικαιοσύνη. Όλα αυτά θα πρέπει ήδη από το 2013 να ξεκινήσουν και έχουμε ένα όραμα που εκθέτει ο Επίτροπος Πίμπαρξ πάνω σε τρεις πυλώνες στους οποίους εδράζεται. Να επικαιροποιηθούν και να εξυγχρονιστούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας. Να υπάρξει μια δέσμη τέτοιων στόχων που θα διασφαλίζει ελάχιστα επίπεδα διαβίωσης κάτω από τα οποία δεν, πρέπει κανείς να αφήνεται να φυτοζωεί. Αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας πυλώνας. Δεύτερος πυλώνας, επικέντρωση στις θέσεις απασχόλησης, εργασίας, ισοδίκαιο πεδίο δράσης, ευκαιρίες, δικαιοσύνη, δικαιώματα του ανθρώπου. Και εδώ η πίστη του είναι ότι χωρίς την, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα παραμείνει η φτώχεια. Λοιπόν η αξιοπρέπεια είναι ο πυρήνας του δεύτερου πυλώνα. Και ο τρίτος πυλώνας είναι σαφές ότι πρέπει να είναι η βιωσιμότητα, η αηφορία. Υπάρχει ισχυρή διασύνδεση με τη συζήτηση για τη συνέχεια follow από το Ρίο μετά από 20 χρόνια για την ε, διατήρηση ε, και διασφάλιση των ε, στόχων για την αηφορία ορατά όλα αυτά σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές ορατά και έχουν επιπτώσεις και στη φτώχεια και στον αγώνα που δίνουμε για την καταπολέμηση αυτής της κατάστασης της φτώχειας. Και μετά προφανώς έχουμε και την πρόκληση της εκρίζωσης της φτώχειας που πρέπει να εντάσσεται μέσα στο πρίσμα του αυξανόμενου πληθυσμού των ε, ανθρώπων που ζουν στην οικουμένη σε αυτόν τον πλανήτη. Από 7 σε 9 δις θα αυξηθούν ε, οι άνθρωποι σε αυτόν τον ε, πλανήτη και θα πρέπει να λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη αυτήν την αύξηση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική και γι' αυτό και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, χωρίς μια καλή διαχείριση και διακυβέρνηση όσον αφορά τους φυσικούς πόρους, το φυσικό πλούτο, αυτά όλα θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις τάσεις όσον αφορά τη μάχη, τον αγώνα που δίνουμε για την καταπολέμηση της φτώχειας. Το ανέφερα ήδη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Επίτροπο Πίμπαλξ, ότι στη διεργασία συζήτηση των μελλοντικών αναπτυξιακών στόχων ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται σε καταστάσεις ευάλωτων κρατών και καταστάσεων και σειράξεων. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους γεγονότα σε πάρα πολύ φτωχές και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Και τι άλλο, για να είμαστε πιο ακριβή και ακριβοδίκαιο. Ο επίτροπο Πίμπαξ θεωρεί ότι πρέπει να επικεντρώσουμε το έργο μα σε τρει στόχου ε, όσον αφορά του ευάλωτου ανθρώπου, ε, ευάλωτου πολίτε. Πρώτα απ' όλα του πιο φτωχού, Δεύτερον, τι γυναίκε που συνεχίζουν να υφίστανται τι επιπτώσεις της αρνητικής μεταχείριση. και εκείνου που ζουν σε απομακρυσμένε περιοχέ και που δεν έχουν τι ευκαιρίε που έχουν άλλοι σε αυτή τη μάχη κατά τη φτώχεια. Σε αυτά τα, ε, τα σε αυτά τα σημεία πρέπει να εδραστούμε στην, ε, ε, στη μάχη που δίνουμε και να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους στόχους. Από τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους εμπλεκόμενους, ένας αριθμός σημαντικών ε, σκέψεων και συμπερασμάτων απορρέουν. Πρώτο από όλα αυτά είναι ότι υπάρχει διαδεδομένη αίσθηση η εντύπωση που έχουν αποκομίσει κάποιοι ότι οι ορισμοί για τους ε, αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας του 2002 καθορίστηκαν ιδιαίτερα από την επιρροή των χορηγών, της κοινότητας των χορηγών και πολλοί λένε ότι αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο αυτό το πλαίσιο κατά κάποιο τρόπο οδήγησε στο να έχουμε μια παραδοσιακή φιλανθρωπιστικού φιλανθρωπικού χαρακτήρα προσέγγιση που αφήνει τις χώρες αυτές να συνεχίζουν να εξαρτώνται από τους ε, ευεργέτες εντός εισαγωγικών χορηγούς. Πρέπει πιο σφαιρικά να προσεγγίσουμε αυτή την προσπάθεια να διασφαλίσουμε μεγαλύτερα πλαίσια συμμετοχής από τις ε, χώρες εταίρους από πλευράς μας και η ομάδα υψηλών αξιωματούχων ε, θέλει να διασφαλίσει ότι οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων εταίρων θα πρέπει να αντανακλώνται και θα πρέπει αυτοί να επομίζονται το έργο με τις απόψεις τους για την ανάπτυξη. Να λάβουμε υπόψη ότι όλες οι προσπάθειες για την ανάπτυξη που πρέπει να κινητοποιήσουμε, οι χώρες αυτές θα πρέπει να, ε, που επομίζονται αυτό το βάρος θα πρέπει να συμμετέχουν για τον καθορισμό αυτής της νέας προσέγγισης στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Δεύτερον, οι εμπλεκόμενοι λένε ότι χρειάζεται ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την αμοιβαία λογοδοσία και αυτό πρέπει πάλι να εξεταστεί ιδιαίτερα εξειδικευμένα και συγκεκριμένα για την αναζήτηση ενός νέου πλαισίου για την αναπτυξιακή προσπάθεια. Πώς θα διασφαλίζεται αμοιβαία η λογοδοσία και από πλευρά των χορηγών και από πλευρά των αναπτυσσόμενων χωρών εταίρων από την άλλη πλευρά. Και τέλος, ως κατακλείδα υπάρχει μια ιδέα που παρουσιάζεται, αναφύεται αυτή τη στιγμή. Ακόμα και καθορίζοντας σφαιρικούς παγκόσμιους στόχους πρέπει να προβλέψουμε κάποια ελαστικότητα και μια προσέγγιση που θα επιτρέπει στις χώρες εταίρους να προσαρμόζουν αυτή την προσέγγιση στις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Η ισοπεδωτική προσέγγιση κοινή προσπάθειας για όλους είναι κάτι καλό ως ε, βιτρίνα ή κάτι το οποίο ω επίφαση μπορεί να λειτουργεί αλλά πρέπει οι εταίροι εκείνοι οι οποίοι οι ίδιοι εμπλέκονται να καθορίζουν αυτές τις ανάγκες και τις προσαρμογές που χρειάζονται μέσα σε αυτό το σφαιρικό πλαίσιο. Τώρα καθώς ξεκινά αυτό το έργο ο Επίτροπος Πίμπαλξ ε, θέλει ιδιαίτερα, επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ρόλο πρωτοπόρου, προπομπού σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι από κοινού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο και κράτη-μέλη, να μπορούμε να είμαστε ηγετικοί και προσωπικότητες και ηγετικά θεσμικά όργανα σε αυτή την προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση που θα μπορέσουμε να προασπίσουμε στο περίγυρο με τις χώρες εταίρους και στο επίπεδο του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτήν ακριβώς τη στιγμή ολοκληρώνει μια πρώτη ανακοίνωση η οποία καθορίζει και συμπεριλαμβάνει τις γενικότερες αρχές που προτείνουμε για μια τέτοια προσέγγιση από πλευρά της ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ανακοίνωση θα αφορά και θα αναφέρει αναφέρεται σε δύο θέματα. Για πρώτη φορά σε ένα κείμενο την αναπτυξιακή ε, ημερήσια διάταξη ως θεματολόγιο και τη συνέχεια που θα δοθεί σε αυτή την προσπάθεια μετά το 2015 για την ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι οι δύο αυτοί στόχοι, ο καθορισμός της ε, βιώσιμης αυτής προσέγγισης για την ε, ανάπτυξη ως ατραπό, ως ε, πορεία και για τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, πρέπει σε μια αμφίδρομη τέτοια προσπάθεια να καθοριστεί. Αναμένουμε ότι αυτό το έγγραφο αυτής της ανακοίνωσης θα ολοκληρωθεί κατά το Φεβρουάριο. Θα παρουσιαστεί κατά τα τέλη Φεβρουαρίου και σίγουρα ο Επίτροπος Πίμπαλξ θα ήθελε ιδιαίτερα να προσέλθει και να παρουσιάσει αυτό το έγγραφο, αυτό το έντυπο στο Ευρωκοινοβούλιο εφόσον θα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προηγούμενα μετά την έγκρισή του. Επιπρόσθετα σε αυτή την ανακοίνωση όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα τελευταία δύο έτη υπό την ηγεσία του Επιτρόπου Πίμπαλξ έχει συντάξει διάφορα έγγραφα τα οποία θα συνεισφέρουν σε αυτή τη συζήτηση. Ανακοίνωση για την υγεία, ένα από αυτά. Ένα για την κοινωνική προστασία ένα άλλο για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Το θεματολόγιο της ημερήσιας διάταξης για τις αλλαγές, αλλά θέματα φορολόγησης επίσης ε, στις ε, χώρες εταίρους. Και με όλα αυτά τα κείμενα θεωρούμε ότι προετοιμαζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί με ιδιαίτερα θετικό τρόπο για να ξεκινήσει η συζήτηση για μετά το 2015 όσο αφορά το πλαίσιο για την ανάπτυξη. Θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό φυσικά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητηθούν αυτέ οι ιδέες μα με το Ευρωκοινοβούλιο, με του ευρωβουλευτέ. Και όπως είπα αυτό το ανέφερα, επιθυμεί ιδιαίτερα σφόδρα ο Επίτροπος Πίμπαξ να προσέθει και να συζητήσει αυτές τις ιδέες μας μαζί σας. Και θα δούμε από κοινού αν με τον Επίτροπο Ποτότσνη θα μπορούσε να γίνει αυτό που είναι και συνυπεύθυνο για αυτή τη διάσταση της ανακοίνωση τη Επιτροπής από πλευρά μα. Περιμένουμε λοιπόν να προχωρήσει η συζήτηση. Ελπίζουμε να μπορέσουμε κάποια από τις βασικές αρχές που σας παρουσίασα να μπορέσουμε να αντισυζητήσουμε την παρουσία και του ιδίου του Πίμπαλξ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ιδέες αυτές εκ μέρους του Επιτρόπου πριν δώσω το λόγο στη Ρεμπέκα Γκρίνσπανγκ να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι επιτυχής θα πρέπει να ακούγεται με μία φωνή και θα πρέπει να είμαστε όχι απλοί οι παρατηρητές της συναντήσεις κορυφής αλλά πρωτοπόροι στις προτάσεις. Έχουν γίνει ε, ε, σημαντικά επιτυχή βήματα και θα πρέπει να ανταλάβουμε υπόψη μας όπως και τα αποτυχημένα βήματα. Ε, τρία τελευταία σημεία έχουμε μείνει πίσω στους στόχους για την υγεία και αυτοί θα πρέπει να ξαναγίνουν προτεραιότητα και βάζω εδώ και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα τα οποία είναι αναπόσπαστο τμήμα του κομματιού που αφορά τους στόχους στον τομέα της υγείας και της υγιεινής. Θα ήθελα να μεταφέρετε λοιπόν προς τον κύριο Πίπαλξ ότι σας υποστηρίζει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το σημαντικό θέμα. Ταυτόχρονα θα ήθελα να υπογραμμίσω και την σημασία που θα έχει ένας ισχυρός πολιτικός διάλογος, στον οποίο θα εμπλέκονται όλοι οι, σε αυτή τη φάση ενδιαφερόμενοι, διασφαλίζοντας την βασική θέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται να μην αγνοήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για το πλαίσιο του 2015. Έλλειψη διακρίσεων είτε με βάση την ηλικία, τον φιλετικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, το φίλο φυσικά, επιμένουμε στο φίλο και στην ταυτότητα του φίλου ιδιαίτερος. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο στην βοηθό Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την κυρία Γκρινσπάιν. Δεν χρειάζεται να την παρουσιάσει κανείς, αλλά φυσικά θα την παρουσιάσω. Είναι στην Επιτροπή Ανοικοδόμησης των Ηνωμένων Εθνών και ήταν εκπρόσωπος και του Μπιλ Κλίντον σε διάφορα ε, φόρα υψηλού επίπεδου. Πριν εργαστεί για τα Ηνωμένα Έθνη ήταν αντιπρόεδρος στην Κωνσταντίνα από το 1994 μέχρι το 1998. Ήταν επίσης Υπουργός Κατοικίας, ήταν Υπουργός Συντονισμού, ήταν Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρος α, γενικά. Έχει ασχοληθεί με το θέμα της μείωσης των ανισοτήτων, της δημιουργίας της κοινωνικής συνοχής και της βελτίωσης της θέσης των γυναικών. Η κυρία Γκρίνσπαν έχει πάρα πολλά να προσφέρει σε σχέση με τις εμπειρίες της, σε σχέση με τα μαθήματα τα οποία όλοι έχουμε πάρει και σε σχέση με τις προκλήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας. Έχετε το λόγο κυρία Γκρίντσπαν. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και για την πρόσκλησή σας, είναι μεγάλη τιμή για μένα και χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση να επαναλάβω κάποια θέματα τα οποία έχουν ήδη υποθεί, αλλά τα οποία νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Έχω τέσσερα μηνύματα να στείλω. Καταρχάς, να σας πω ε, περί τίνος πρόκειται. Το πρώτο μου μήνυμα, όπως είπαν και άλλοι, είναι ότι οι στόχοι αυτοί ε, μας έχουν επιτρέψει να κάνουμε βήματα πρόοδου, όχι γιατί θα πετύχουμε όλους τους στόχους, αλλά ε, και υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στις χώρες, αλλά έχουν υπάρξει βήματα επιτυχή. Και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν είναι ακόμα πεπισμένοι για τη χρησιμότητα των στόχων αυτών. Πολλοί πιστεύουν ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει και τίποτα δεν γίνεται και πρέπει εκεί που έχουν υπάρξει βήματα θετικά να υπογραμμιστούν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ήδη έχουμε διαπιστώσει ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε σε σχέση με το 2015. Έχουμε τρία χρόνια ακόμα ε, σήμερα τα πράγματα πάνε καλά, αλλά μέσα σε τρία χρόνια μπορεί, αν χάσουμε γενικά ε, το μήνυμα, να αποτύχουμε. Το τρίτο μήνυμα. Έχουμε πολλά να μάθουμε επίσης ε, και από τη μία και από την άλλη. Βλέπουμε ποια ήταν τα άσχημα πράγματα που κάναμε, βλέπουμε ποια είναι τα κενά τα οποία έχουμε μπροστά μας. Και βλέπουμε το τι έχουμε κάνει καλά και μία τελική σκέψη αν θέλετε σε σχέση με τους κινδύνους που υπάρχουν. Υπάρχουν κίνδυνοι, δεν υπάρχουν εγγυήσει σε σχέση ε, με το πώς θα πάνε τα πράγματα με το πλαίσιο μετά το 2015. Να πω τώρα γιατί έχουμε κάνει θετικά βήματα μέχρι τώρα, πώς το πετύχαμε αυτό. Δεν θα επαναλάβω όλους τους αριθμούς, γιατί έχουν υποθεί με σωστό τρόπο θα έλεγα. Δύο διαφορετικά πράγματα όμως τα οποία πρέπει να υπογραμμίσω. Πρώτον, οι στόχοι αυτοί και τα προγράμματα μας πέτυχαν επιτρέποντας την λειτουργία ενός πλαισίου ε, που επιτρέπει την ανθρώπινη ανάπτυξη, κρατώντας πάντα ε, σε ε, περίοπτη θέση θα έλεγα ε, το πρόσωπο ε, αυτών οι οποίοι ωφελούνται. Ανατομέα φυσικά και αυτό το ανθρώπινο ιδιαίτερα χαρακτηριστικό θα πρέπει να διατηρηθεί και για την ατζέντα μετά το 2015. Θα πρέπει να συνδεθούν οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και ένας από τους δείκτες τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαζί με τη διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι οι τάσεις για τις μειώσεις αναστράφηκαν από το 2008. Σε σχέση με τα ODA υπήρχε μια πτωτική τάση μετά το 2008, μετά όμως από τις δηλώσεις για τους στόχους της χιλιετίας τα πράγματα αναστράφησαν. Δεύτερον, να πούμε ότι υπήρξαν επιτυχείς ε, ε, προτάσεις από πλευράς των κυβερνήσεων. Πρέπει να ξέρετε ότι σε 60 χώρες οι στόχοι εσωτερικεύθηκαν, εντάχθηκαν ε, και στις δημοσιονομικές προοπτικές και στο δημοσιονομικό πλαίσιο των ιδίων των κρατών. Και αυτό είναι σημαντικό. Ένα, τρίτο, ένα τρίτο στοιχείο στο οποίο πρέπει να υπογραμμίσω είναι το ότι έχουν κάνει τα NPGs για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών δόθηκαν νέα μέσα στην κοινωνία των πολιτών να προωθήσουν κάποιες στόχους και ιδέες ε, και για να προωθήσουν ένα επικοδομητικό διάλογο με τις κυβερνήσεις και ένα ε, μέσο για να παραμείνουν οι κυβερνήσεις υπόλογες, να μπορούν να ελέγχονται οι κυβερνήσεις από πλευράς της κοινωνίας των πολιτών. Η σημασία αυτού του μέσου είναι κάτι το οποίο είχε παραγνωριστεί μέχρι τώρα και είναι θα έλεγα ένας από τους βασικούς λόγους για τα επιτυχή βήματα που έχουν γίνει σε σχέση με τα MTGs. Ένα στοιχείο λοιπόν το οποίο θα ήθελα να σας αφήσω σαν δείκτη είναι ότι 370 εκθέσεις προόδου έχουν γίνει αντικείμενο παραγωγής σε εθνικό επίπεδο, όχι για τις διεθνείς εκθέσεις, όχι για τις σφαιρικές εκθέσεις, όχι για τις περιφερειακές εκθέσεις. Εγώ μιλάω για εθνικό αυστηρά επίπεδο. 370 εκθέσεις προόδου έχουν συνταχθεί ε, και σε σχέση με την δράση ε, της κοινωνίας των πολιτών και σε σχέση με την δράση των κυβερνήσεων και σε σχέση με τον διάλογο ανάμεσα στους δύο. Τώρα, σχετικά με τους στόχους, τους ίδιους στόχους. Όπως είπαμε, υπάρχουν ορισμένοι στόχοι οι οποίοι έχουν ε, ε, επιτευχθεί, δεν θα τους επαναλάβω. Παρ' όλα αυτά, όταν ε, μιλάμε ότι προσπαθήσαμε να κόψουμε στα δύο την ακραία μορφή ένδυας, και πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το πετύχαμε κυρίως σε σχέση με την Κίνα ή και μέσω της Κίνας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πράγματι η Κίνα ήταν ένας πρωταγωνιστής σε σχέση με τη μείωση κατά 50% της ακραίας ένδυας. Αλλά υπήρξε πρόοδος και σε άλλες χώρες τις οποίες δεν συζητάμε. Και ακόμα και στην υποσαχαρική Αφρική. Έχει, υπήρχε έλλειψη προόδου μέχρι το 2010 περίπου θα πρέπει επίσης και στην υπόλοιπη Νοτιοανατολική Ασία να δούμε ότι υπήρξαν εφετικά βήματα σε σχέση με την καταπολέμηση της ένδυας και όχι μόνο στην Κίνα. Η επίτευξη λοιπόν των στόχων σε σχέση με τον τομέα της υγείας τώρα. Εδώ θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε ότι οι μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν σε σφαιρικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικοί, καθοριστική σημασίας. Να προσθέσω εδώ αυτό σε σχέση με αυτά που μας έδωσε σαν στοιχεία ο κύριος Τέιλορ. Έχουμε 40% μείωση της, της ε, θνησιμότητας στην φυματίωση, 30% αντίστοιχα στην ελονοσία και οι νέες λοιμώξεις έχουν μειωθεί κατά 25 με 30%. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποτρέψει 2,5 εκατομμύρια θανάτων. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, τώρα Ας πάω γρήγορα τώρα στο δεύτερο μήνυμα που θέλω να στείλω ε, στο ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η πορεία προς την πρόοδο. Δεν θα πρέπει να ε, εφησυχάσουμε. Η πρόοδος θα πρέπει να γίνει αντικείμενο επιτάχυνσης από το 2015 και μετά έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό αποτυχίας επίτευξης των στόχων. Συνεπώς πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά για το 2015 και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβραδύνουμε τις προσπάθειες. Αν επιβραδύνουμε τώρα, τα επόμενα τρία χρόνια θα τα χάσουμε και το 2015 δεν θα αναφερόμαστε στους στόχους σαν μια επιτυχή εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. οι βασικοί στόχοι στους οποίους έχουμε μείνει πίσω είναι η, παιδική, η μητρική θνησιμότητα και η παιδική θνησιμότητα, κυρίως όμως η θνησιμότητα των μητέρων. Έχουμε μείνει πίσω και στο περιβάλλον, έχουμε μείνει πίσω επίσης και στη συνεργασία σε επίπεδο περιφερειακό και σφαιρικό. Θα ήθελα εδώ να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη σημασία και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων. Αναγνωρίζεται αυτή η προσπάθεια από το σύνολο των Ηνωμένων Εθνών και σε 44 χώρες έχουν δημιουργηθεί νέα προγράμματα και νέα στήριξη για την επίτευξη όλων των στόχων στους οποίους έχει υπάρξει η σε επίπεδο εθνικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας ε, των ε, μητέρων, στον τομέα της εξυγίανσης ε, των υδάτινων πόρων, εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Ένα τρίτο μήνυμα σχετικά με το τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο η ηγεσία από πλευράς των κυβερνήσεων και η ε, αίσθηση ιδιοκτησίας των προγραμμάτων από πλευράς της κοινωνίας. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί. Όπως είπα και όπως είπε προηγουμένως και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα να ξεχωρίσουμε τις διαφορές ανάμεσα σε χώρες έτσι ώστε οι συγκεκριμένες αυτές προσπάθειες επίτευξης των στόχων να γίνουν με τον καλύτερο κατά περίπτωση τρόπο. Ε, να πω επίσης ότι μέσω της προσπάθειας επίτευξης των στόχων έχουμε και το θέμα του μοχλού, του πολλαπλασιαστή από την προσπάθεια αυτή. Μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα και παράλληλα και πρέπει να προχωρήσουμε με αυτή την παράλληλη πορεία. Τρίτον, η ισότητα των φύλων έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την επίτευξη όλων των στόχων και όχι μόνο σε επίπεδο γενικών στόχων. Ξέρουμε ότι έχει μεγάλη σημασία το θέμα των φύλων και παρόλα αυτά εκεί που μένουμε πίσω, επαναλαμβάνω, είναι η λεγόμενη ε, μητρική θνησιμότητα και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει άμεση σχέση με την αποκατάσταση της ισορροπίας των φύλων. Ε, επίσης, το θέμα της κοινωνικής προστασίας έχει πάρα πολύ σημασία αυτό για τη συνολικότερη πρόοδο. Η πρόοδος δεν μπορεί να είναι βιώσιμη εφόσον δεν καλύψουμε τους πληθυσμούς από τις ανάγκες ε, της συγκυρίας και από τα εξωτερικά σοκ. Πρέπει να μην ξεχνάμε και την τοπική και περιφερειακή διάσταση και την παρέμβαση των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, όχι μόνο το εθνικό επίπεδο και το διεθνές φυσικά. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει το πλαίσιο αμοιβαία ευθύνη με παράλληλη αξιολόγηση και εποπτεία και με πραγματικές εθνικές συμμαχίες. Τρία πράγματα τώρα, τα οποία στα πλαίσια της προσπάθειας των στόχων πρέπει να υπογραμμίζουμε τρία πράγματα ε, στα οποία δεν πήγαμε καλά και πρέπει να τα διορθώσουμε για το πλαίσιο μετά το 2015. Πρώτον, υπάρχει το ότι οι χώρες οι οποίες στάθηκαν ικανές να σημειώσουν σημαντικότατη πρόοδο, χρησιμοποίησαν τα ODAs, αλλά δεν έχουν την δυνατότητα να τα αντικαταστήσουν και για τον ιδιωτικό τομέα, για να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα σε εσωτερικό επίπεδο. Τα ODA παραμένουν σημαντικά, αλλά για να μπορέσουμε να κλιμακώσουμε προς το καλύτερο την κατάσταση, απαιτείται κινητοποίηση σε εθνικό επίπεδο και αύξηση του ποσοστού των ιδιωτικών επενδύσεων. Εκεί δεν πήγαμε καλά. Το δεύτερο σημείο στο οποίο δεν πήγαμε καλά είναι οι διακρίσεις και οι ανισότητες οι στατιστικές δεν αναφέρονται σωστά στους εύθραυστους πληθυσμούς. Οι μέσοι όροι δεν καλύπτουν τους εύθραυστους πληθυσμούς. Όπως λέμε και στην ισπανική γλώσσα, θα πρέπει να ξεφύγουμε από την δικτατορία των μέσων όρων, γιατί οι ευάλωτοι πληθυσμοί δεν αντικατοπτρίζονται στους μέσους όρους. Και τέλος, για να κλείνω. Η προσπάθεια που έγινε ήταν εκ των άνω. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σήμερα με την εκ των άνω προσπάθεια. Να πω ότι ήδη από τώρα έχουν υπάρξει 100 χώρες οι οποίες έχουν υποσχεθεί και δεσμευθεί για εθνικές διαβουλεύσεις στο επίπεδο αυτό. Και εμείς καλύπτουμε τις 50 μόνο. Οι υπόλοιπες 50 γίνονται από τις ίδιες τις χώρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο θα υπάρξουν 11 θεματικές διαβουλεύσεις για όλα τα θέματα και θα υπάρξει και μια σφαιρική ιονή διαβούλευση για την εμπλοκή των πολιτών μέσω των κοινωνικών μέσων επικοινωνίας. Έτσι θα συμπληρώσουμε λοιπόν τις προσπάθειες και του πάνελ υψηλού επίπεδου και των διοργανικών υπηρεσιών ε, των Ηνωμένων Αθνών και έτσι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε για την επίτευξη των στόχων και για μετά το 2015. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης αργότερα να μπορώσω να σας δώσω κάποιες ε, ιδέες που έχω σχετικά με τους κινδύνους ενός πλαισίου το οποίο να είναι φορτωμένο σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ε, θα πρέπει να υπάρξει κατά κάποιο τρόπο ένας χαρακτηρισμός προτεραιοτήτων εδώ και να επιλέξουμε στόχους οι οποίοι να είναι εφικτοί στην επίτευξή τους και να βοηθήσουν συνολικά τον πρόεδρο, την πρόοδο. Και το άλλο είναι η σύγκληση των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης με, τις, με τα νέα πλαίσια συνεργασίας και θα ήθελα εδώ ε, να μας πει ε, ακριβώς τι γνώμη έχει για τα θέματα της προώθησης της βιωσιμότητας και επίσης ε, του νέου πλαισίου μετά το 2015. Thank you very much, Rebecca, for Ευχαριστώ πολύ τη Ρεμπέκα για αυτή την τόσο σημαντική συνεισφορά της. Δίνω λίγο περισσότερο λόγο στου ομιλητέ, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε και κατόπιν θα κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Έχω την τιμή να καλωσορίσω και να δώσω το λόγο στον κύριο Βιταλή Μέγια, ο οποίο συντονιστή του ε, δικτύου Reality of Aid, που είναι ένα δέκτυο ε, αφρικανικό για να υπερασπίσει την ε, εκρίζωση της ένδυας και είναι και μέλος της Διευθυντικής Επιτροπής ε, της Εκστρατείας για τους ε, Στόχους των Ανθρώπων. Θα συμφωνείτε κι εσείς ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική και συνολική αναπτυξιακή πολιτική και γι' αυτό δίνω ιδιαίτερα χαρά το λόγο στον κύριο Μέγια για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είναι τιμή για μένα να είμαι προσκεκλημένος εδώ ως ομιλητής ε, στο πάνελ αυτό. Όπως βλέπετε, ευθύς εξ αρχής ε, ότι εμάς μας δίνετε 10 λεπτά και δίνετε στους υπολείπους 15 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Θα συνεχίσω από αυτά που είπε η συνάδελφος που μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία της. Για μας, από την αφρικανική πλευρά, είναι ανάμεικτες οι αντιδράσεις όσον αφορά τους ε, στόχους της χιλιετίας. Καταρχάς, ε, η Ήπειρος έχει ακόμα το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων ε, που βιώνουν με απόλυτη φτώχεια, απόλυτη ένδια. Επομένως για μας οι στόχοι της χιλιετίας είναι ακόμα πρόκληση και οι περισσότερες από τις κυβερνήσεις προσπαθούν να δουν πώς μπορούν να βελτιώσουν τα διάφορα μοντέλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιτύχουν τους στόχους μέχρι το 2015. Πέραν αυτού όμως, υπάρχουν και κάποια διδάγματα. Καταρχάς, η παγκόσμια οικονομική σταθερότητα είναι ζωτική σημασία για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Πριν από την ε, οικονομική κρίση, η Αφρική τα πήγαινε πολύ καλά και μάλιστα μπορούσαμε να επενευόμαστε και ότι είχαμε σχεδόν επιτύχει το στόχο του να μειώσουμε την ε, ένδια στο μισό της. Αλλά μετά από την κρίση όλη η πρόοδος η οποία επετεύχθη σιγά σιγά αρχίζει να εξαφανίζεται και εν μέρει αυτό γίνεται λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Λόγω της κρίσης δεν μπορούμε να λάβουμε μεγαλύτερη ενίσχυση για την επίτευξη των στόχων και επίσης οι αγορές για τα προϊόντα μας έχουν μειωθεί έχουν συρρυκνωθεί και επομένως είναι τεράστια πρόκληση για τις κυβερνήσει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τους στόχους της χιλιετίας. Δεύτερον, η προσέγγιση εκ των άνων ε, στην οποία αναφέρθηκε η συνάδελφος δεν έχει αποτελέσματα στην πραγματικότητα, διότι δεν περιλαμβάνει όλους αυτούς οι οποίοι επηρεάζονται απευθείας. Ε, οι κυβερνήσεις κατασκευάζουν σχολεία, νοσοκομεία, μιλάτε για αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αναφέρεται κανείς στους δασκάλους που θα διδάξουν σε αυτά τα σχολεία, τους γιατρούς που θα δουλέψουν σε αυτά τα νοσοκομεία, πώς θα τους πληρώσουμε. Δεν αντιμετωπίζει κανείς αυτά τα θέματα. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία εάν τα παραμερίσουμε θα ε, επηρεάσουν ιδιαίτερα την επίτευξη της πρόοδου που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Και μάλιστα οι ίδιοι πολίτες αναρωτιούνται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι επινόησαν αυτούς τους στους στόχους της, ε, της χιλιετίας και πώς αντιμετωπίζουν οι στόχοι αυτοί τις ανάγκες που έχω εγώ στο χωριό μου. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο για τους τεχνοκράτε να τα πλουστεύσουν όλα αυτά σε ένα χωριό και να καταλάβουν για παράδειγμα ότι η αλληλεία κατά κάποιο τρόπο είναι αυτή η οποία θα φέρει ψωμί στο τραπέζι στο τέλος της μέρας. Επίσης μάθαμε ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα είναι βασικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Και γιατί το λέω αυτό. Πριν από την τελευταία χρονιά, η Λιβύη, την Ισία και κάποιες άλλες χώρες της περιοχής ε, θεωρήθηκαν ε, απτά παραδείγματα για τις υπόλοιπες χώρες της υποσεχάριας Αφρικής ε, και θα έπρεπε και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας. Επειδή όμως οι πολίτες δεν συμμετέχουν απαραίτητο στα προγράμματα αυτά, συμβαίνει το εξής έχουμε τη σταθερότητα η οποία όμως στην πραγματικότητα ε, καταστρέφει όλα τα προγράμματα τα οποία έχουμε εξελίξει. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ειρήνη εάν θέλουμε να επιταχύνουμε τους στόχους της χιλιοτίας. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι το γεγονός ότι οι στόχοι της χιλιετίας για χώρες οι οποίες τις έχουν εντάξει στα εθνικά τους προγράμματα ε, δίνουν αποτελέσματα. Επομένως, αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αναπτυξιακά σχέδια χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των στόχων της χιλιετίας διαπιστώνουμε ότι έχουν συντονισμό, προγραμματίζουν το πότε θα έχουν αποτελέσματα και προσαρμόζουν και τον προπολογισμό τους ώστε να λάβουν υπόψη το θέμα αυτό. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι της χιλιοετίας έχουν συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό για τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού, της ποιότητας των αποτελεσμάτων προς τους πολίτες επιτόπου, αλλά επιπλέον υπάρχει και αυτό το στοιχείο της ιδιοκτησίας, ότι κάπως αυτή η στόχη της χιλιετίας είναι δική μας και οι πολίτες έχουν ταυτιστεί με αυτούς. Αλλά επίσης να σας πω ότι διαπιστώσαμε και κάτι καινούριο μέσω των στόχων της χιλιετίας οι κυβερνήσεις πλέον μπορούν να επενδύσουν περισσότερο σε μέσα κοινωνικής προστασίας. Μπορούν να προσφέρουν ενισχύσεις στους αγρότες επιτόπου. Μπορούν να επενδύσουν περισσότερα σε νοσοκομεία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν στο παρελθόν λόγω του μακροοικονομικού πλαισίου που τους είχε επιβληθεί. Αλλά επειδή ε, οι στόχοι της χιλιετίας τους δίνουν την ελευθερία να το κάνουν αυτό, σε κάποιο βαθμό βλέπουμε ότι οι κυβερνήσεις αρχίζουν να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομής και ε, κατάλληλες θεσμικές ε, ε, μορφές που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους πολίτες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μαλάουι. Πριν από 10 χρόνια περίμενε ε, επιστημιστική βοήθεια κάθε χρόνο. Ε, η κυβέρνηση κατόπιν αποφάσισε όμως ότι η επιστητική βοήθεια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν άμεσα και επομένως γιατί αυτό είναι απειλή και έτσι άρχισε να επιδοτείται και τώρα το Μαλάουι είναι καθαρός εξαγωγέας αραβοσίτου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δόθηκε η όθηση από πλευράς κυβέρνηση για να εξετάσουν νέους καινοτόμου τρόπους να επενδύσουν και να δημιουργήσει αυτό και εισόδημα. Κάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της εσωτερικής κινητοποίησης των πόρων. Νομίζω ότι σιγά σιγά ε, αυξάνεται η εσωτερική κινητοποίηση πόρων και οι κυβερνήσεις το χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες που έχουν στον προπολογισμό τους. Αυτό όμως θα πρέπει να συμπληρωθεί και από εξωτερικούς πόρους και εξωτερική χρηματοδότηση. Εμείς μάλιστα λέμε ότι μας, υποσχεθήκατε 0,7% περισσότερο και εξακολουθούμε να μην λαμβάνουμε αυτά τα κονδύλια και μας φέρνει και σε δύσκολη θέση να το συζητάμε. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι εμείς βελτιώνουμε και ενισχύουμε την εσωτερική κινητοποίηση πόρων και θέλουμε να δούμε και άλλη προσπάθεια, διότι πρόκειται για σύμπραξη, εταιρική σχέση. Θέλουμε να δούμε λοιπόν προσπάθεια και από τους εταίρους μας σε αναπτυξιακό επίπεδο για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους με την παρούσα κρίση η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια μάλλον θα μειωθεί. Αλλά εμείς λέμε ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Αν θέλουμε να επιταχύνουμε την επίτευξη των στόχων της χιλετίας μέχρι το 2015, δεν θα πρέπει να σταματήσουμε, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να αντιμετωπίσουμε τα κενά τα οποία διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή. Πέραν όμως του 2015, εμείς ως κοινωνία αυτό το οποίο έχει σημασία να κάνουμε είναι να σκεφτούμε χωρίς στεγανά και να δούμε τι έχει σημασία για τους πολίτες, ώστε να μην είναι απλώς ένα αμάλγαμα διαφόρων πολιτικών που ο καθένας θα πρέπει να επιτύχει, να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ιδέες, ιδέες οι οποίες θα προέλθουν από τους πολίτες και αυτά όλα να τα μεταμορφώσουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα έχει αποτελέσματα. Και το θέμα της δημοκρατικής ιδιοκτησίας των απτυξιακών προγραμμάτων είναι σημαντικό, διότι μόνο έτσι θα προέρθουν ιδέες από τους πολίτες, θα συμμετέχουν οι πολίτες στο σχεδιασμό και θα δεσμευθούν σε θέματα ε, λογοδοσίας, παρακολούθησης και ούτω καθεξής. Διότι εάν απουσιάζουν οι πολίτες θα είναι πολύ δύσκολο να ζητήσουν ε, ευθύνε από την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν είναι το πιο σημαντικό. Αλλά πρωτίστως, ιδίω για τους φτωχούς αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε είναι πώς θα αυξηθεί η πρόσβαση και ο έλεγχος των παραγωγικών μας πόρων διότι έχουν κουραστεί όλοι ε, με όλη αυτή την ε, ε, υπόθεση της, ε, της φιλανθρωπίας. Το 75% των κατοίκων της Αφρικής θεωρεί ότι το 2015 θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Αφού λοιπόν έχει αλλάξει η νοοτροπία, θα πρέπει πλέον να εντάξουμε τους πολίτες στο επίκεντρο της ανάπτυξης. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και πώς θα εκδημοκρατιστεί το κράτος και οι κοινωνικοί θεσμοί που δίνουν, προσφέρουν υπηρεσίες στους ανθρώπους. Και για μας αυτές είναι μία από τις βασικές πτυχές τις οποίες θα πρέπει να εξετάσουμε, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να είναι και σημαντικοί παράγοντες οι πολίτες. Εάν λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε πέραν του 2015, θα πρέπει να ε, αναπτύξουμε την προσέγγιση που θα βασίζεται στον άνθρωπο. Για μας αυτό είναι υψής της σημασίας. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε και να εγκρίνουμε πολιτικές και νόμους και να έχουμε τους μέγιστους δυνατούς πόρους για να προωθήσουμε και να εκμεταλλευτούμε πλήρως τα πολιτικά ε, και πολιτιστικά δικαιώματα. Αυτά αποτελούν το κλειδί της πρόοδου. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε και κάποια στοιχεία των στόχων της χιλιετίας, κυρίως το θέμα της ένδυας και της ανισότητας. Και για μας αυτό έχει μόνο αποτέλεσμα εάν εξετάσουμε πώς θα γίνει ανακατανομή των φόρων, πώς θα βελτιώσουμε τις δημόσιες δαπάνες για τις κοινωνικές πολιτικές και πώς θα ενισχύσουμε τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας και τα κοινωνικά προγράμματα τα οποία φορούν απευθεία στους πολίτες. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό ε, το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας για τους πολίτες. Πρέπει να δούμε πώς θα τους δώσουμε πρόσβαση σε πολιτιστικές υπηρεσίες αλλά και πρόσβαση σε γη και σε όλες τις ε, υπηρεσίες που χρειάζονται για να την εκμεταλλευτούν. Ένα λεπτό παραπάνω, δύο λεπτά παραπάνω μου δώστε, ένα μου έμεινε. Νομίζω τα ίδια θέματα συζητούμε κι εμείς, αλλά θεωρούμε ότι πρωτίστως πρέπει να ε, συζητήσουμε τα θέματα της ε, κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας από πλευράς περιβάλλοντος και πώς θα τα εντάξουμε όλα αυτά στο όλο πλαίσιο. Το πιο σημαντικό, κύριε Πρόεδρε, είναι και το θέμα της καλής διακυβέρνησης, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς θα ενισχύσουμε τη συμμετοχή των πιο ευάλωτων ε, φορέων στου παγκόσμιου θεσμούς πώς θα ε, εντάξουμε τη συμμετοχή των πολιτών σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Μόνο από αυτή τη βάση μπορούμε να συζητήσουμε θέματα ιδιοκτησία, κύριε Πρόεδρε. Και τέλο, υπάρχει το θέμα του πώ μπορούμε να προχωρήσουμε και πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ιδέε για μετά το 2015. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια ε, συλλογική προσπάθεια που θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερομένους για να καταλήξουμε σε αυτές τις ιδέες. Ε, ώστε σε κάθε πάνελ, σε κάθε πλαίσιο που χρησιμοποιείται να υπάρχει κάποιο στοιχείο συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών αλλά και των υπολείπων ενδιαφερομένων ώστε να έχουμε συνολικά αυτό το νέο παγκόσμιο πλαίσιο. Να μην έχουμε μόνο κρατική ιδιοκτησία, αλλά δημοκρατική ιδιοκτησία, στην οποία οι πολίτες και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μέρ. Καθώς ξεκινήσαμε με κάποια καθυστέρηση, θα επεκτείνω, θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε στις 11 και 5, αλλά θα παρατείνουμε με τη συμφωνία του κύριου Κατσμάρακ μέχρι τις 11 ε, και 10. Ο κύριος Γκέρενς είπε ότι ήθελε να λάβει τον λόγο μετά η κυρία Ντεκεζέρ. Παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Σας ευχαριστώ. Mr. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει μέρος στις μεγάλες αυτές συνδιασκέψεις σχετικά με τους στόχους της χιλιετίας υπάρχουν δύο τμήματα. Ε, υπάρχει το υπουργικό κομμάτι και εκεί βαριούνται όλοι γιατί όλοι λένε τις ίδιες ιστορίες, τις ίδιες στατιστικές και τις ίδιες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, τις οποίες συνήθως δεν ε, σέβονται ή σέβονται εν μέρη. και για λόγους πολιτικής ορθότητας ε, δεν λέμε την αλήθεια. Και μετά έχετε την κοινωνία των πολιτών η οποία συνεδριάζει. Εκεί πράγματι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Πολλές φορές υπάρχουν και ψευδεστήσεις βέβαια θα πρέπει νομίζω ότι το πολιτικό κομμάτι να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρον. Ένα δεύτερο θέμα, να προσπαθήσουμε να βρούμε τις ευθύνες όλων των εταίρων. Έχετε φτωχού στη ΣΥΠΑ, στην Κίνα, στο Μαλάουι. Η πρώτη χώρα είναι μια αναπτυγμένη χώρα, όπου η εσωτερική αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι η απάντηση στη φτώχεια. Είναι μια απάντηση η οποία δεν αναλαμβάνεται πλήρως. Έχετε φτωχού στην Κίνα η Κίνα δημιουργεί πλούτο, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και φτώχεια. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν θα πρέπει απλά να διαπιστώνουμε ότι έχουν κρυζώσει ένα τμήμα της φτώχειας, θα έπρεπε να τα καταφέρουν καλύτερα, όπως και όλες οι αναδυόμενες χώρες. Και μετά έχετε μια τρίτη χώρα σαν το Μαλάουι, που είναι υπό ανάπτυξη χώρες η οποία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να τα βγάλει πέρα. Εκεί πρέπει να αναλάβουμε εμεί τις ευθύνες μας, δεν έχουμε πετύχει τους στόχους μας πλήρως. Θα πρέπει να δράσουμε και να προσπαθήσουμε να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες από τη μία και την άλλη πλευρά. Να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Εσείς, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε κάνει την επιλογή της διαφοροποίησης και σας στηρίξαμε πολιτικά σε αυτό. Δεν θα πρέπει να τεθεί να αμφισβητήσει συγκεκριμένη επιλογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη έχει προτείνει την λεγόμενη ε, συμπεριληπτική ή ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις επιλογές της. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις αυτές να επηρεαστούν ακόμα περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι μέχρι σήμερα. Ο Μάικελ ε, μου δείχνει ότι πρέπει να σεβαστώ το χρόνο. Είμαι σκεπτικός πάντως κλείνω σε σχέση με το τι έχουμε πετύχει. Δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν θα πρέπει βέβαια να είμαστε και μονίμως παραπονούμενοι. Θα σκάνουμε λοιπόν κάποιες προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης. Κινδυνεύουμε να κολλήσουμε σε μια συζήτηση στρατοσφαιρικού τύπου, μακράν της πραγματικότητας. Έχω κι άλλα να σας πω, αλλά δυστυχώς δεν έχω χρόνο. Μπορώ να ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι σύντομοι, γιατί έχουμε σε λίγη ώρα να ξεκινήσουμε το επόμενο κομμάτι της συζήτησης. Η κυρία Ντοκεζέρ έχει το λόγο. κάποια σημεία σε σχέση με αυτά τα οποία υπόθηκαν μέχρι τώρα. Και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο Σάρλα. Είναι αλήθεια ότι προχωράμε σε περιόδους δημοσιονομικής ε, λιτότητας και ε, σε σχέση με τον ετήσιο προϋπολογισμό και σε σχέση με το πολιετές πλαίσιο. Γνωρίζουμε ότι η βοήθεια γενικά στον τομέα της ανάπτυξης ε, θα περιοριστεί, για να μην πω σε κάποιες περιοχές θα περικοπεί σοβαρά. Εξαρτάται λοιπόν τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε με τους στόχους ε, της χιλιετίας, γιατί προβλήματα θα δημιουργηθούν. Και θα συμφωνήσω εδώ με αυτά που έλεγε ο Σάρλα. Τι ρόλο παίζει η πολιτική ηγεσία σε όλα αυτά. Εγώ εκπλήσωμαι στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας, σαν παράδειγμα, βλέποντας ότι πράγματι ταυτίζουμε βάζουμε στον ίδιο σάκο χώρες οι οποίες είναι δυνητικά πλούσιοι φυσικοί πόροι, είναι εξαιρετικά σημαντικές και ξέρετε ότι στην υποσαχαρική Αφρική υπάρχουν τέτοιες χώρες, όπου το κλίμα δεν είναι κλίμα ε, πραγματικής ε, ξηρασίας, όπου όμως ε, η παιδική θνησιμότητα είναι ενδυμική τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο πολιτικό με αυτές τις κυβερνήσεις, πώς μπορεί να πιέσει και ποιοι είναι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων μπορούμε είτε απλά να ασκήσουμε πιέσεις, είτε να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει περαιτέρω κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά σε καμία περίπτωση θα μας πούν οι κυβερνήσεις δεν θα πάμε εμείς να δώσουμε λεφτά στις χώρες που έχουν τα μεγαλύτερα χρυσορυχεία. Ναι, είναι λίγο υπεραπλουστευμένη η απάντηση αυτή. Πρέπει να διαφοροποιηθεί η στάση μας απέναντι στις χώρες οι οποίες δεν έχουν πόρους και σε αυτές που έχουν πόρους. Για μας λοιπόν σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να διαφοροποιήσουμε την πολιτική μας απάντηση. Αν δεν το κάνουμε δεν θα είμαστε αξιόπιστοι σε καμία περίπτωση. Νόιζερ και μετά η κυρία Θεοχάρου σα ευχαριστώ πολύ Μάικλ. Δύο πολύ σύντομε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς την εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Αφενός γνωρίζετε είμαι μεγάλος υπέρμαχο ώστε εμεί στου αναπτυξιακού στόχου της χιλιετία μετά το 2015 την πρόσβαση στην ενέργεια να, να το καταστήσουμε ω θέμα σε έναν αυθύπαρκτο στόχο της ε, ανάπτυξης ε, για του στόχου χιλιετία. Χωρί αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Πώ έχουν τα πράγματα. Ξέρω ότι ο επίτροπο Πίμπαξ δραστηριοποιείται και προ την ε, κατεύθυνση αυτή έχει αναλάβει και κάποιε πρωτοβουλίε. Τι γίνεται. Δεύτερη ερώτηση προ τον ΟΗΕ. Κάνατε λόγο μόλι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ομιλεί με μία φωνή. Με μία φωνή να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη. Υπάρχει όμω τώρα μία προσέγγιση σε τριγωνική και σχέσει να εργαζόμαστε. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά κράτη από κοινού κράτη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση σε τριγωνικέ σχέσει θα εργάζεται για το μέλλον τη συνεργασία. Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία παράδειγμα. Δανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία. Ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα τέτοια προσέγγιση. Ποια είναι η δική σας αντίδραση και αντιμετώπιση αυτής της πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Σε ευχαριστώ πολύ κυρία Θεοχάρους, ε, παρακαλώ να είσαστε σύντομοι όλοι, θα είναι πραγματικά επικοδομητικό. Ευχαριστώ, κυρία Θεοχάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μπορούσε να με είχε καλύψει κανείς περισσότερο από τον κύριο Μέια, ο οποίος έθεσε νομίζω τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση και δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας ή στην στρατόσφαιρα, όπως είπε ο κύριος Γκέρνς είναι πολύ σημαντικό να εγγύψουμε στις πραγματικές ανάγκες των φτωχών σε όλο τον πλανήτη και όχι να προσπαθούμε μέσα από ένα ευρωπαϊκό ε, γίγνεσθε το οποίο δεν επιτρέπει σε καμιά περίπτωση να πούμε ότι μπορούμε να εξαγάγουμε δημοκρατία ή να εξαγάγουμε καλές πρακτικές. Ας δούμε πρώτα την άθλια κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να προσπαθούμε να ε, διορθώσουμε τους άλλους πρέπει να τονίσουμε την στήριξή μας στη δέσμευση για 20% της αναπτυξιακής βοήθειας όσον αφορά την υγεία και την παιδεία. Το έχει θέσει πάρα πολύ σωστά ο κύριος ε, Μέγια γιατί αν δεν έχουμε δασκάλους, αν δεν έχουμε γιατρούς, αν δεν έχουμε νοσηλευτές που να παραμένουν στον τόπο τους δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε καμία δημοκρατική, καμία κοινωνία, όχι μόνο δημοκρατική κοινωνία. Και θα ήθελα τη δέσμευση και των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν ότι θα παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό το θέμα, στην, στο, σε, αυτή την στόχευση. Τώρα, όσον αφορά το νέο πλαίσιο, ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οπωσδήποτε θα ε, στηρίζεται στο ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της χιλιετίας το 2015. Εκεί είναι πάρα πολύ ασαφές το ζητούμενο. Και εφόσον μιλήσαμε για την παιδεία, όσον αφορά την υγεία, ε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχουμε και τη διαβεβαίωση ότι ε, οργανώσεις όπως το Global Fund, για παράδειγμα, το οποίο έχει αποδεδειγμένα εργαστεί με ζήλο και αποτελεσματικότητα στον τομέα της αντιμετώπισης της μαλάριας, του AIDS, της φυματίωσης, ε, και στην επίδευξη των στόχων 4, 5 και ειδικά του στόχου 6 ε, θα εξακολουθήσει να στηρίζεται ισχυρά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την ε, Κομισιόν πρωτίστω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελένη, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ Ελένη. Και ο κύριος Κορτές παρακαλώ, τελευταίος. Σας ευχαριστώ, δεν έχουμε χρόνο αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι μια σύντομη περίληψη κάποιων από τα θέματα που θα ήθελα να αναπτύξω περισσότερο. Πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε μπροστά από, μία, από μία από τις μεγαλύτερες ιδέες που υπήρχαν για την ανθρωπότητα, για τους στόχους αυτούς ε, της χιλιετίας για την ανάπτυξη οικουμενική δέσμευση για την εκρίζωση της φτώχειας. Εξάπαντος, ε, οικουμενική δέσμευση όλων προς ένα κοινό στόχο. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε μια τέτοια ιδέα. 15 χρόνια πέρασαν, 12-13 χρόνια και λείπουν ακόμα 2 χρόνια και δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να προαγάγουμε κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ετών ώστε αυτά τα οποία έχουν ε, επιτευχθεί ήδη να είναι το δυνατόν τα βέλτιστα, τα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Δεύτερον, θα ήθελα να υπογραμμίσω επίση και τη συμμετοχή, όπω είπε ο κύριος Μέγερ θέλουμε σε σχέση με την ανάπτυξη για τους στόχους χιλιετίας να αυξηθεί αυτό σε σχέση με τις αναψώμενες χώρες. Πρέπει να λάβουμε πάρα πολύ υπόψη αυτές τις ανάγκες αυτών των χωρών και να συμμετάσχουν αυτές πλήρως. Μια άλλη ιδέα σε σχέση με την κυρία Greenspan. Είπε ότι θα υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση ανοιχτή για την κοινωνία, όλη η κοινωνία των πολιτών να συμμετάσχει για, την ανάπτυ... για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Μια οικουμενική τέτοια πρωτοβουλία μπορούμε και τα κοινοβούλια να χρησιμοποιήσουμε, τα εθνικά κοινοβούλια ως σημείο αναφορά, ώστε από τα εθνικά κοινοβούλια επίση να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε επαφέ με όλε τι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις ΜΚΟ και να διευρύνουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το δίκτυο, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή, ώστε η τελική συμφωνία να είναι πιο οικουμενική, η πιο σφαιρική που θα γίνεται και να ικανοποιηθούν το δυνατόν περισσότεροι και να ευθυγραμμιστούν όλοι για την εκρίζωση τη φτώχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω απλά τον λόγο στην κυρία Γκρίνσπαν. Ένα λεπτό για να απαντήσει. Με το χρονόμετρο θα σταματήσουμε και μετά ο κύριος Μάγερ, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν. Αν κατάλαβα καλά την παρέμβασή σας, την ερώτησή σας, για τις ε, ε, ευρωπαϊκές χώρες, σε τριγωνικές ε, τέτοιες συνεργασίες βλέπουμε ότι έχουμε 30 σε σχέση με την ανοιχτή ομάδα για την ε, πρόοδο για τους ε, στόχους χιλιετίας. Όλοι θέλουν να συμμετάσχουν και πρέπει να έχουμε ομαδικές κατηγοριοποιήσεις, ας το πω έτσι, δυνατότητες συνεργασίας, ώστε περισσότερες χώρες να μπορούν να συμμετάσχουν. Αυτό δεν διαφέρει από άλλα θεσμικά όργανα, ε, για παράδειγμα, όπου θα πρέπει να έχουμε ε, για παράδειγμα κάποιον που είναι πρόεδρος ή προεδρεύων και μια, άλλη, ε, μια ομάδα χωρών που συμμετέχουν και συνοδεύουν ως συμπρόεδροι αυτές τις δραστηριότητες. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Για τα κοινοβούλια είχαμε και μια συνάντηση στο κήτο του σημερινού του Εκουαδόρ ε, που το Μάρτιο προβλέπεται να διεξαχθεί και ελπίζω ότι θα υπάρξει η εμβάθυνση στην συμμετοχή των κοινοβουλίων σε αυτή τη διαδικασία μέσα στο πλαίσιο του μετά το 2015. Ευχαριστώ πολύ Ρεμπέκα. Και ο κύριος ε, Μάιερ έδειξε ότι δεν χρειάζεται να παρέμβει. Εξαιρετικό αυτό και μπορούμε να ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να λάβει υπόψη αυτά τα θέματα. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε όσους παρενέβησαν και μπορώ να δώσω τώρα τον λόγο στο δεύτερο πάνελ. Στον αξιότιμο κύριο Κατσμάρεκ που θα είναι ο πρώτος ε, που θα ηγηθεί του δεύτερου πάνελ. Ο κύριος Κατσμάρεκ, καλή σας μέρα. Το δεύτερο πάνελ θα δει το δυναμικό και την δυνατότητα δράσης για το πλαίσιο του μετά το 2015 και να δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να συνεχίσει να εμπλέκεται σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι πραγματική χαρά να είμαι πρόεδρος σε αυτό το πάνελ, να προεδρεύω ως εισηγητή για αυτό το ιδιαίτερα προκλητικό θέμα, ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα και πιστέψε με δεν είναι καθόλου εύκολο το εγχείρημα αυτό. Είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά υπάρχουν τόσε πολλέ εναλλακτικέ δυνατότητε, τόσε πολλέ ιδέε. Είναι τόσο πολύ σύνθετο το θέμα και περίπλοκο που είμαι ευγνώμων που έχουμε αυτή την ακρόαση σήμερα. Για μένα είναι μεγαλύτερη ευκαιρία να ακούσω, να αφούγκραστώ τι απόψει σα και να σημειώσω και να τι λάβω υπόψη ω παρατηρήσει και σχόλια ερωτήματα και τα λοιπά για να συνεχίσω τη δουλειά μου. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο ε, Πέδρο Μορασάν ε, και να τον ευχαριστήσω αυτόν από το Ίδρυμά του και την ομάδα του, τον κύριο Άρνο Μπέκρεν, την κυρία Μόνικα Αλέση και τον Γιάννους ε, για την εκπόνηση αυτής της μελέτης με τον ίδιο ακριβώς τίτλο και λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς τα μελήματα και τις ανησυχίες της δημόσιας αυτής ακρόασης. Δίνω τον λόγο στον δόκτωρα Μορασάν αμέσως στη συνέχεια. Παρακαλώ κύριε Μορασάν. Λειτουργεί το μικρόφωνο, μάλιστα. Θα κάνω την παρουσίαση αυτή στα ισπανικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πρόσκληση αυτή να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης μας. Σε πολλές πτυχές δεν υπάρχουν αντιφάσεις, ε, θεμελιώδεις αντιφάσεις ή ε, αντιρρήσεις για όσα εκφράστηκαν. Υπάρχει υψηλό βαθμός συνένεση. Έτσι λοιπόν, πολύ γοργά από πλευρά μου, για μια συνεισφορά σε αυτή τη συζήτηση, θα εργαστούμε σε τέσσερα θέματα ω άξονε ουσιαστικά, που είναι αυτά τα θέματα που συμπεριλαμβάνει η μελέτη. Πράγματι, το πρώτο τμήμα είναι μια εισαγωγή και η έκθεση του οράματος. Ποιοι είναι οι στόχοι της ε, ανάπτυξης για τη χιλιετία, η αναπτυξιακή στόχη χιλιετίας. Δεύτερον, μετά το 2015 ποια είναι η διαδικασία και η διεργασία, ποιο είναι το πλαίσιο για την ανάπτυξη που αναζητούμε να πετύχουμε. Το τρίτο είναι πολύ σημαντικό ω άξονα. Με ποιο τρόπο θεωρούμε εμεί ότι η δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πιο ενδυναμωμένη, πιο ενισχυμένη. Και με βάση όλε αυτέ τι τρει πτυχέ κάνουμε κάποιες συστάσεις που συντάσουμε, Καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα και κάνουμε τις συστάσεις μας. Λοιπόν, χωρίς αμφιβολία, και συμφωνούμε με την κυρία Ρεμπέκα Γκρίνσπαν επ' αυτού, χωρίς αμφιβολία οι στόχοι της χιλιετίας, αναπτυξιακή αυτή στόχη στέφθηκαν με επιτυχία. Ήταν μια επιτυχία σε πολλές πτυχές, υπό πολλέ συνιστώσει και έδωσαν έντονη πρόθεση στην ε, διεθνή οικονομική συνεργασία, δεσμεύοντα αυτή τη συνεργασία σε μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένους δίκτες και εξειδικευμένου ε, δείκτε. Αυτό είναι το πιο ισχυρό χαρτί αυτής της ε, προσπάθεια. Συνένεση σε παγκόσμιο επίπεδο και που σε σχέση με άλλες πλευρές για την διεθνή πολιτική λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πτυχές η αναπτυξιακή στόχη της χιλιετίας είναι σαφής είναι λειτουργικοί και μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Όπως μπορείτε να δείτε στο γράφημα, η διαδικασία αυτή ήταν πολύ διαφοροποιημένη και η επίτευξη των στόχων της ηλιετίας ήταν πολύ, ε, η επίτευξη ήταν πολύ διαφορετική. Δεν θα επισέλθουμε σε αυτό, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό το γεγονός. Ωστόσο, πέρα από αυτά πρέπει να δεχθούμε ότι θέλοντας να δούμε προς το μέλλον τι θα κάνουμε και εδώ πάλι υπάρχουν ευάλωτα ε, στοιχεία. Αφενός δεν υπάρχει μία ε, διαφοροποιημένη προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τις ε, γεωγραφικές διαφορές όσον αφορά το ζήτημα της ανάπτυξης. Γι' αυτό η επιτυχία στην καταπολέμηση της φτώχειας βασίζεται ουσιαστικά όπως αναφέρθηκε για παράδειγμα για την Κίνα. Ενώ αλλού σε άλλα μέρη του κόσμου έχει εγγραφεί ως μήμα της ημερήσιας διάταξης στο θεματολόγιο. Απ' την άλλη πλευρά η κυβερνητικές οργανώσεις δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους νέους, ε, τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος και που πλήττονται όχι μόνο οι φτωχές χώρες αλλά σήμερα ακόμα και οι αναπτυσσόμενες χώρες. Αρκεί να δούμε τις ειδήσει ε, σε παγκόσμιο επίπεδο για να δούμε για ποιο πράγμα κάνουμε λόγο και να καταλάβουμε αυτή την εξέλιξη. Υπό το δικό μας πρίσμα πρέπει να πούμε ότι καταδεικνύουμε και λέμε ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να πάει πιο πέρα, ακόμα πιο πέρα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τεράστια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν μπροστά τους. Και Λαμβάνοντα υπόψη τι διαφορέ και αντιθέσει που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, το μόνο διεθνέ ε, όργανο διακυβέρνηση που μπορεί να υπομειστεί αυτό το ρόλο, ηγετικό ρόλο στον, στην κατάρτιση και σχεδιασμό μια ημερήσια διάταξη μετά το 2005 για την ανάπτυξη είναι τα Ηνωμένα Έθνη, λαμβάνοντα υπόψη και τα όσα δεσμευθήκαμε να πράξουμε στο παρελθόν. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε τις ε, ε, τάσει που αυτή τη στιγμή διαγράφονται παράλληλα με παράλληλη εξέλιξη. Αφενός έχουμε την θέσπιση του High Level Panel της ομάδας υψηλών αξιωματούχων τον Ιούλιο 2012. Αφετέρου από την άλλη πλευρά είδαμε ότι αυτό το πάνελ είχε δύο συναντήσεις. Μία συνεδρίαση στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και η επόμενη συνάντηση στην ε, Ινδονησία ώστε μετά το Σεπτέμβριο εφέτος να έχουμε ένα, μια ειδική εκδήλωση των Ηνωμένων Εθνών όπου θα παρουσιαστεί αυτή η έκθεση της ομάδας υψηλών αξιωματούχων High Level Panel. Προχώρησε η συζήτηση για το θεματολόγιο μετά το 2015. Έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις και η έκθεση της ομάδας εργασίας συμπεριλαμβάνει τα θέματα που ανέφερε ο κύριος Μέγερ. Μια approach, μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα δικαιώματα του ανθρώπου και μια άλλη διάσταση που είναι η ανάπτυξη, που οι πτυχέ τη ανάπτυξη, ξεχωριστέ πτυχέ που πρέπει να εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο όμω δεν έχουμε την ίδια δυναμική με τη διαδικασία μετά το 2015 ελπίζουμε ότι θα υπάρξει επιτάχυνση των πραγμάτων για να μπορούμε να κάνουμε λόγο πραγματικά ότι και οι δύο αυτές διεργασίες θα μπορούν ε, αμφίδρομα να ε, δίνουν ερεθίσματα και ε, κίνητρα η μία στην άλλη. Πρέπει να συγχαρούμε τα Ηνωμένα Έθνη ώστε με αφορμή αυτό το γεγονός τουλάχιστον καταβάλλεται προσπάθεια τώρα να έχουμε μια διαδικασία που θα είναι bottom-up, εκ των κάτω προς τα πάνω. Και γι' αυτό σε αυτή τη διαργασία με τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις δύο ειδών. Οι διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο, μια ομάδα χωρών που ε, καλύπτεται από αυτές τις διαβουλεύσεις, κυρίως ε, φτωχότερες χώρες, αλλά επίσης έχουμε τις θεματολογικές διαβουλεύσεις αυτή η διαδικασία είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό το Ευρωκοινοβούλιο να το γνωρίζει αυτό για να μπορεί να συναγάγει τα αναγκαία συμπεράσματα και να δράσει σωστά. Και ιδιαίτερα επειδή εργαζόμαστε ενάντια στο χρόνο, ενάντια στο χρονόμετρο, λαμβάνοντα υπόψη ότι θα έχουμε μια ειδική εκδήλωση το Σεπτέμβριο ήδη. Δηλαδή υπάρχει μια διεργασία, μια θεσμική διεργασία με άλλα λόγια, στην οποία συνδυάζονται οι διεργασίες, ας το πω έτσι, διαβούλευσης στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών, στο επίπεδο των κοινοβουλίων, στο επίπεδο των χωρών, των κρατών μας, με θεματολογικές διαβουλεύσεις για τα θέματα που προανέφερα. Αλλά Όμως επίσης, υπάρχουν... άλλη πλευρά και κάτι άλλο. Υπάρχει μια συζήτηση που λαμβάνει υπόψη τις διεργασίες ε, που ε, έγιναν προηγούμενα. Για παράδειγμα, 20 χρόνια μετά το Ρίο Ντεζανέιρο το αστέρι αυτό, ας το πω έτσι, το πιο λαμπρό στον ορίζοντα όσον αφορά συμφωνίες για την ανάπτυξη δεν μπορεί να αγνοηθεί. Καταφέραμε στο τέλος με ένα κείμενο που πολύ γοργά διατυπώθηκε να απαριθμίσουμε επιλεγμένα 24 θεματολογικά πεδία που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και να εντάσσονται όταν εξετάζουμε τη δυνατότητα δέσμευσης ε, των ε, ε, αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τις δράσεις μας. Με βάση όλες αυτές τις διεργασίες θεωρούμε ότι η συζήτηση δεν είναι ακαδημαϊκού πανεπιστημιακού χαρακτήρα και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το οποίο αποκαλούνται τρεις εναλλακτικέ δυνατότητες που θα είναι πολύ σημαντικές για τη συζήτηση. Πρώτη, να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους κοινούς στόχους αλλάζοντας ε, μόνο κάπως τους δείκτες που υπάρχουν για τη χρήση αυτή για το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ε, μέχρι το 2025 σε ένα χρόνο ορίζοντα. Η άλλη δυνατότητα που υπάρχει είναι να επεκτείνουμε κατά κάποιο τρόπο, με σημαντικό τρόπο, το πλαίσιο αυτό ως ένα ε, επαυξημένο πλαίσιο που θα συμπεριλαμβάνει συνενετικά πεδία μέσα στη διεργασία αυτό. Ωστόσο αυτό ως είναι γνωστό είναι λίγο πιο επίμαχο θέμα. Υπάρχει και μια τρίτη εναλλακτική λύση που θεωρούν οι συντάκτες ότι θα ήταν η ιδανική, η καλύτερη. Οι προκλήσεις για την ανθρωπότητα, αυτό το οποίο αποκαλείται το πλαίσιο ή στρατηγική, στρατηγική ενός οικουμενικού ενιαίου κόσμου. One World που με ένα γράφημα το οποίο αντανακλά την πρόταση αυτή. Αυτές είναι οι τρεις ε, σημαντικότερες εναλλακτικές προτάσεις για τη συζήτηση σε σχέση και με το Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ έχουμε τις ιδέες αυτών των τριών τύπων στρατηγικής, αυτών των τριών διαφοροποιημένων διεργασιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, δείκτες που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη, θεσμικά όργανα που θα μπορούν να συμμετάσχουν. Είναι μια περίληψη βέβαια. Φυσικά υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ λύσεις που δεν είναι ευκταίες και που για τη δική μας κρίση δεν είναι ε, λειτουργικές και αποτελεσματικές. Να ολοκληρωθούν όλα αυτά το 2015 και να μην ξεκινήσει τίποτα το καινούριο. Θεωρούμε ότι πολιτικά όχι κάτι τέτοιο θα ήταν μόνο ανεύθυνο, αλλά ήταν, είναι πραγματικά κάτι επικίνδυνο υπάρχει μια ελάχιστη συνένεση και με βάση αυτή τη συνένεση πρέπει να εργαστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, είναι μια προσπάθεια να δούμε πώς αυτά τα 25 θεματολογικά πεδία ή επίπεδα μπορούν να ενταχθούν σε μια κοινή διαργασία, να υπαχθούν σε αυτήν για την αηφορία στην ανάπτυξη υπό τις διάφορες συνιστώσεις, τις τους. Κοινωνική, οικονομική, ε, βιώσιμη προοπτική. Η προσπάθεια προσπάθεια να ενταχθούν όλα αυτά μέσα στην προοπτική Ρίο μετά από 20 χρόνια. Για να κάνουμε λόγο για τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο πράγματα. Πρώτον, ποια ήταν ποια ήταν η προσπάθεια που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιτυχία της. Δεύτερον, ποια είναι τα δυναμικά, ποιο είναι το δυναμικό και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν βασικά θεμελιώδη έγγραφα που αναφέρθηκαν εδώ και που λαμβάνονται υπόψη, υπόψη ως μια βάση, κοινή βάση για τη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε το θεματολόγιο για την μεταμόρφωση ε, σε σχέση με το 2015, όπου βρίσκεται και το στοιχείο της ε, ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Έχουμε επίσης τη δημόσια διαβούλευση που προσανατολίζεται προς μια ημερήσια διάταξη μετά το 2015, ε, ήδη το καλοκαίρι του 2012. Έχουμε τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις του Συμβουλίου, έχουμε τη μελέτη που εκπονούμε τώρα εμείς ε, για αυτούς τους στόχους και στο τέλος τέλος θα έχουμε και την έκθεση που θα συντάξει η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, του Ευρωκοινοβουλίου Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τα έγγραφα είναι τα θεμελιώδη έγγραφα και έντυπα για να πετύχουμε μια ημερήσια διάταξη στην προσπάθειά μας που θα ενεργοποιήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξεκινά από μηδενικό σημείο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα από του μεγαλύτερου, ε, ε, α το κινητήρες ε, σε αυτή την προσπάθεια και ο μεγαλύτερο χορηγό σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν κατάφερε όμω να υλοποιήσει αυτέ τι υποσχέσει και πρέπει να το δεχθούμε αυτό, ώστε να επιτευχθεί το 0,7% του ΑΕΠ για του στόχου για την ανάπτυξη. Και αν τα δούμε στατιστικά όλα αυτά, η βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση ευτυχώς δεν ε, υπέστη σημαντικές διακοιμάσεις ή μειώσεις παρόλη την οικονομική κρίση. Είναι όμως σημαντικό να διατηρηθούν οι προσπάθειες για να διασφαλιστεί αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας. Πρέπει να προαχθεί περισσότερο η διεργασία συνοχής και συνεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πολύ καλά παρουσιάζεται να προαχθούν τα, οι κοινοί στόχοι. Είναι τεράστια πρόκληση που μπορεί να διαδραματίσει διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ ένα πολύ σημαντικό ρόλο ανταποκρινόμενη στο ρόλο που πρέπει να υπομειστεί. Ο πιο σημαντικός ωστόσο ρόλος στην πρόκληση αυτή είναι ο θεσμικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμπληρωματικότητα, η παραπληρωματικότητα σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συμπλήρωμα και των κρατών μελών και των προσπαθειών τους. Γι' αυτό οι προκλήσεις είναι τρεις ουσιαστικά. Πρώτον, να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερα αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί και που υπήρξαν θετικές συνεισφορές ε, για τους στόχους αυτούς, να υλοποιηθούν οι διεθνείς συμφωνίες για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας του θεματολογίου ε, του, της Συμφωνίας των Παρισίων και αυτή η προαγωγή να τύχει να προαχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να είμαστε πολύ πιο φιλόδοξοι. Αυτό είναι η δεύτερη παρατήρηση παρατήρηση, στη εταιρική σχέση για την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει να παίρνουμε περισσότερο στα σοβαρά την πολιτική συνοχή και να έχουμε μεγαλύτερη δέσμευση όσον αφορά τα θέματα ε, στο παγκόσμιο επίπεδο ε, του παγκόσμιου πλούτου. Και το 0,7% που πρέπει να μπορέσει να προωθηθεί και να βελτιωθεί για να κερδίσουμε τη χαμένη αξιοπιστία κάπως. Αυτές οι συστάσεις λοιπόν με άλλα λόγια είναι αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει να απευθύνουν μια έκκληση, έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπέρ όλης της προσπάθειας για τη διαβούλευση αυτών των θεμάτων. Λαμβάνουμε υπόψη την πείρα που συνελέγει σε σχέση με όλη αυτή την προσπάθεια. Στη μελέτη εμείς εκινούμε από το σημείο ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα πολύ σημαντικό κοινοβούλιο σε διεθνές επίπεδο. Είναι ένα σημαντικό κοινοβούλιο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι ένα κοινοβούλιο ίσως ακόμα πιο σημαντικό. Ένα από τα τρία πιο σημαντικά στοιχεία για αυτή τη διεργασία. Γι' αυτό το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να υπομειστεί ένα ρόλο ας το πω έτσι, σημαντικό για να διασφαλιστεί η επιτυχία μετά το 2015 των στόχων, αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Γι' αυτό προτείνουμε να είναι πιο δραστηριοποιημένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιο ενεργό ρόλο να αναλάβει. Τα εξή τέσσερα επόμενα σημεία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά. Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να καταβάλει τεράστια προσπάθεια ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια κοινή ενιαία θέση, σαφή κοινή ενιαία θέση και ισχυρή θέση μέσω μιας έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου που θα δίνει καλύτερη προώθηση και με πιο αποτελεσματικό τρόπο της ε, Διεθνούς ημερήσιας Διάταξης για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας προς την ανάπτυξη μετά το 2015. Δύο, το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να συναγάγει τα συμπεράσματα από την πείρα που έχει συλλέξει σε παγκόσμιο επίπεδο για τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις σε σχέση με μια πράσινη οικονομία. Είναι αναγκαία μεγαλύτερη διπλωματική προσπάθεια που θα καταβάλλεται και εσωτερικά στο επίπεδο των κρατών μελών, αλλά και εξωτερικά, ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος και να εμπλακούμε σε ένα διάλογο όχι μόνο με τις πιο φτωχές χώρες της Αφρικής, Ασίας και Λατινικής Αμερικής, αλλά επίσης και ιδιαίτερα με τις αναδυόμενες χώρες, όπως τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα, που διαδραματίζουν ένα πολιτικό ρόλο πάρα πολύ σημαντικό στην ε, ομάδα των 27. Αλλά όχι να επιβάλλουμε μια ημερήσια διάταξη που θα έχουμε εμείς εκπονήσει οι ίδιοι, σε σχέση με αυτές τις χώρες, αλλά να τονίσουμε τις πιο σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να έχει μια ξεχωριστή ε, στεγανή μερίσια διάταξη, αλλά σε συζήτηση με αυτές τις χώρες να υπάρξει μια δυναμική επ' αυτών των διαβουλεύσεων. Χρειάζεται χρόνος εδώ. Έχει μεγάλη ευκαιρία που του προσφέρεται το Ευρωκοινοβούλιο ως κρίκος, κρίκος που συνδέει τα διαφορετικά συμφέροντα και τις διάφορες πλευρές. Σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, για παράδειγμα, η περίπτωση οι θέσεις των πιο περιθωριοποιημένων χωρών που δεν είναι εκείνες που έχουν τον ε, περισσότερο σημαντικό ρόλο και γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε και υποστηρίζουμε το, τη θέση του κυρίου Μέγερ για τις πιο φτωχές χώρες. Θα πρέπει να αναζητήσει στόχους που θα είναι σαφείς το Ευρωκοινοβούλιο, που θα είναι σύντομοι, σαφείς, λειτουργική, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και πιο σφαιρικοί, ας το πω έτσι, πιο ε, ενταξιακή, περισσότερο ενταξιακού χαρακτήρα, ολοκληρωμένου χαρακτήρα, ώστε να δημιουργείται ένα σαφές πλαίσιο συμμετοχής. Να ζητηθεί επίσης να υλοποιηθούν οι οικονομικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα επίπεδα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό είναι ο μόνος ε, τρόπος να κερδίσουμε αξιοπιστία όσον αφορά αυτές τις διαβουλεύσεις. Αξιοπιστία που δυστυχώς είδαμε ότι επλήγει κατά το παρελθόν και σε σχέση φυσικά και με τις ίδιες τις απαιτήσεις που υπήρχαν να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την οικονομική, η χρηματοοικονομική αυτή κρίση. Και πρέπει να δεχθούμε ότι υπάρχουν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν και πολλές προσδοκίες σε σχέση με αυτό το θέμα και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές. Επιμένουμε ότι είναι το πιο σημαντικό όργανο το Ευρωκοινοβούλιο για να